Vamos a empezar la votación. Παρακαλώ, καθίστε για να αρχίσει η ψηφοφορία. Ακούστε με και μια φορά. Yo no te he cogido nada, esto es mío. Hombre, estos son los míos. Bueno, vamos a iniciar el voto. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Έχετε όλοι τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας. Δεν έχει κανένας πρόβλημα, δεν την ξέχασε, όλοι τις έχετε μαζί. Ωραία. Αρχίζουμε την ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε την έκθεση της κυρίας Γκρελιέ για τα τεχνικά μέτρα. Θα θέλετε το λόγο κυρία Γκρελιέ ή μπορούμε να περάσουμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Κατευθείαν. Πολύ ωραία. Ψηφίζουμε κυρία Πατράου Νέβες. Η πρώτη τροπολογία είναι δικιά μου, η δεύτερη είναι του κυρίου Καπόλα Σάντος, αλλά είναι παρομοιότυπες, σχεδόν ταυτόσιμες. Και επειδή θέλουμε να διευκολύνουμε το έργο σας, προτείνουμε συγχώνευση των δύο τροπολογιών. Μία μικρή διόρθωση θέλουμε μόνο και στο σημείο 6-8, στη δεύτερη παράγραφο, να προσθέσουμε 1η Οκτωβρίου 2010, αυτό να το αντικαταστήσουμε από το 31 Δεκεμβρίου 2012, στα σημεία 9.3, 9.6 και 9.8. Μία αλλαγή ημερομηνία. Υπήρξε λάθο εδώ. Αντί να λέμε 1η Δεκάτου 2010, το διορθώνουμε και λέμε 31 Δεκάτου 2012 για τα σημεία 9.3, 9.6 και 9.8. Αυτή η προφορική τροπολογία ισχύει και για τις δύο τροπολογίες, την τρία, τη δική μου και την τέσσερα, του κυρίου Καπόλα Σάντος. Προτείνουμε άλλωστε συγχώνευση των δύο τροπολογιών σε μία ενιαία, γι' αυτό και δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε δύο φορές παρά μόνο μία. Γιατί δεν μας τα είπατε το πρωί όλα αυτά όταν συζητούσαμε τις τροπολογίες, γιατί τώρα διευρύνατε την τροπολογία σας και μας φέρνετε σε δύσκολη θέση. Αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Εντάξει, θα ψηφίσουμε. Εκτός αν έχει κανείς αντίρρηση με την προφορική τροπολογία. Αλλιώς κάνουμε τη συγχώνευση όπως είπατε. Ωραία. Ψηφίζουμε με την διόρθωση την προφορική, μια και δεν αντέδρασε κανείς, τις τροπολογίες 3 και 4 που είναι ταυτόσιμες. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. απορρίπτονται 13 ψήφες κατά. 10 υπέρ, 13 κατά. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1 της ηγητρίας, άρχεται η ψηφοφορία. Σε la votación. Τέλος ψηφοφορίας. Es aprobada por 19 19 ψήφοι υπέρ και 2 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 5 του κυρίου Χάτ, Χάττον. Άρχεται η ψηφοφορία. Se cierra la votación. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 9 ψήφοι πέρα, αλλά 14 κατά. Άρχεται η ψηφοφορία. Διαδικαστικό κύριο Ρωμέβα. Τι συμβαίνει κύριε Ρωμέβα. Η κυρία Λοβίν κατέθεσε συγκεκριμένη προφορική τροπολογία για την ε, δική της τροπολογία 6 Μία πολύ συγκεκριμένη τροπολογία της κυρίας Λέβιν, εκεί που λέει ε, συμμορφώνεται πλήρως, αντί να λέμε το άρθρο, με το άρθρο 13, να διευκρινίσουμε ότι πρόκειται για την παράγραφο 2αβ. Α και Β. Εκεί που λέμε μόνο 13, να λέμε 13αβ. Καλώς. Ψηφίζουμε την τροπολογία 6 με την προφορική προσθήκη. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται με 22 ψήφους κατά. Ψηφίζουμε την τροπολογία 7 του κυρίου Γκάλαχερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Σε Περισσεύει ένας σοσιαλιστής, μια ψήφος παραπάνω. Το μηχάνημα το λέει. Για βρείτε μεταξύ σας. Ε, κάποιος περισσεύει. Περισσεύει μια ψήφος σοσιαλιστών. Επαναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Το μηχάνημα το είπε, δεν φταίω εγώ. Τροπολογία 7 του κυρίου Γκάλεχερ, άρχεται ψηφοφορία. Για να μετρήσουμε πόσοι σοσιαλιστές ψηφίζουν, πόσο το ελέγξουμε αλλιώ. Εκτός αν μπερδεύτηκε και το μηχάνημα, γιατί δεν είναι τέλειο ούτε τα μηχανήματα. Δεν λέω σαν και καλά ότι εσείς φταίτε. Καλώς, το αγνοούμε. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Απορρίπτεται με 14 ψήφους κατά και 9 υπέρ. Τροπολογία 8 του κυρίου Χάττον. Άρχεται η ψηφοφορία. Άρα δεν είναι καλά προγραμματισμένο το μηχάνημα. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 14 κατά 8 υπέρ. Τροπολογία 9 Χάττον. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 8 υπέρ 14 κατά απορρίτεται. Τροπολογία 10 του κύριου Γκάλεχερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Και πάλι 8 υπέρ 14 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 11 του κύριου Γκάλεχερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται ομόφωνα κύριε Γκάλαχερ. Τροπολογία 2, Λέβιν. Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλο Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 4 ψήφους υπέρ και 17 κατά. Και μία αποχή. Ψηφίζουμε τώρα το σύνολο της νομοθετικής πρότασης, όπως έχει τροποποιηθεί, Άρχιτε ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 17 ψήφους υπέρ, 4 κατά και μία αποχή και το σχέδιο νομοθετικού ψηφίσματος τώρα, έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται με 18 ψήφους υπέρ και 4 κατά. Συγχαρητήρια κυρία Γκρελιέ. Τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Συγχαίρω την εισηγήτρια. σε Διάφορα. Υπάρχει τίποτα για τα διάφορα. Όχι. Οπότε το σημείο 13 το διεκπαιρώσαμε. Σημείο 14. Ησυχία παρακαλώ. Ανακοινώσει τη Προέδρου για τις αποφάσεις των συντονισμών. Των συντονιστών, συγγνώμη. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Η στάση των συντονιστών τη 26 η του Μηνό. θα σας έχουν μοιραστεί μέσω τη γραμματείας αν δεν υπάρχουν ε, αντιρρήσει θα θεωρηθούν ως συγκεκριμένες. Οι σημερινές αποφάσεις των συντονιστών θα σας κοινοποιηθούν όσον Η επόμενη συνεδρίασή μας θα γίνει στις Βρυξέλλες 15 και 16 Μαρτίου. Μπορείτε να φύγετε όλοι. Να μείνουν στην αίθουσα παρακαλώ μόνο οι συντονιστές.